προσπάθεια για την εκπόνηση μια στρατηγική εσωτερική ασφάλεια και θα συνεργαστούμε μαζί σα με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση επί του θέματος αυτού. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα την έκθεση Κορνέλης Δε Γιόγκ όσον αφορά την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Για τέσσερα λεπτά το λόγο έχει ε, εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ποινικό δίκαιο δεν είναι ένα θέμα πολύ εύκολο. Αφορά περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπόπτων. Λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Κυρίως χρειάζεται σύνεση όσον αφορά τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα πρέπει να υπάρχουν και καλοί λόγοι για να γίνεται κάτι τέτοιο. Όπως αναφέρεται στα διεθνή μέσα ε, ε, ε, που καθορίζουν και πώς πρέπει να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν ε, να προσέχουμε διότι τα μέσα ενημέρωσης ε, ε, προβάλλουν περισσότερο το έγκλημα σήμερα. Άρα το πολιτικό σύστημα, το δικαστικό σύστημα τελικά οι εισαγγελίες όλοι εκτίθενται. Οι πολιτικοί προσπαθούν να εθετήσουν νέα νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν τις απειλές που δημιουργούνται ή να έχουν μια ευρύτερη νομολογία. Ε, ποια είναι η κεντρική ιδέα. Να πιστούν οι άντρες και οι γυναίκες της Ευρώπης ότι μέσω της θέσπισης νέας νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε μια απάντηση απειλέ που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα. Δεν ισχύει αυτό. Η ιδέα του ποινικού δικαίου δεν είναι οι βραχυπρόθεσμες επιτυχίες. Πριν θεσπιστούν νέοι νόμοι, ή πριν αυξηθούν οι ποινέ, πρέπει να σκεφτεί κανεί πολύ προσεκτικά τι συνέπειε. Στην πραγματικότητα, μπορεί να ελπίσει κανεί ότι θα συλλάβει περισσότερου εγκληματίε και θα του εντάξει καλύτερα στην κοινωνία. Και μακροπρόθεσμα, η κοινή γνώμη πραγματικά ενδιαφέρεται για μεγαλύτερε ποινέ ή απλώς είναι κοινή εντυπωσιασμού για την κοινή γνώμη και ίσως θα μπορούσαν τελικά τέτοια αποτελέσματα επιτευθούν με την υφιστάμενη νομοθεσία. Η άλλη απειλή όσον αφορά το ολοπλαίσιο προέρχεται από τι ε, Βρυξέλλε δυστυχώ. Στι Βρυξέλλε χρησιμοποιούνται μεγάλε εξουσίε ε, που έχουν επεκταθεί έτη περαιτέρω από τι συνθήκε Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Διάφορα ε, έχει υιοθετηθεί κάποια κοινή προσέγγιση όσον αφορά, εναρμόνιση όσον αφορά κάποια ε, ποινικά δικήματα και κάποια μικρότερο, μικρότερα δικήματα εναρμονίζονται όταν χρειάζεται. Λοιπόν, ε, υπάρχουν και άλλα νέα δικήματα, νέα εγκλήματα που χρειάζονται ε, καθορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι καλό να προσπαθούμε να σεβαστούμε τις διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση. όσον αφορά λοιπόν το ποινικό δίκαιο, αναφέρεται ότι αν οι τη Ευρωπαϊκή Ενώση είναι αντίθετε προς το Σύνταγμα μπορούν να κινηθούν διαφορετικά τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν ευρύτερε εξουσίε από τη μία πλευρά και από την άλλη ανάγκη σεβασμού εθνικών παραδόσεων. Άρα αυτά δημιουργούν εντάσει αυτέ οι δύο πτυχέ. Το ποινικό δίκαιο δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί με τον ίδιο τρόπο σε άλλου τομεί, όχι κατακαιρματισμένα. Χρειάζεται συντονισμό, ενιαία προσέγγιση. Αν δεν υπάρξουν πραγματικοί λόγοι για τις αλλαγές δεν πρέπει να γίνονται. Στην έκθεσή μου καθιστώ σαφές ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ποινικό δίκαιο σαν μια ευκαιρία, σαν ένα τομέα, σαν μια αρένα για να κάνουμε επίδειξη διαμόρφωσης πολιτικής. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τη θέμενη αξία η ασδήποτε εναρμόνισης πρέπει να αποδεικνύεται από στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πριν αλλάξει το ποινικό δίκαιο πρέπει να βρούμε άλλες αποτελεσματικότερες λύσεις και θα πρέπει να γίνουν και διάφορε δοκιμέ κατά πόσο είναι αναγκαία η αλλαγή τη νομοθεσία. και θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή, μια συνέπεια. Άρα όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουν τα αναγκαία, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Χρειάζεται συντονισμός. Κατακαιρματισμένο ποινικό δίκαιο δεν είναι καλό. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου, τη Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών για τη τεράστια υποστήριξη που παρήχαν στην εκθεσή μου και στην ομάδα εργασία. Ελπίζω να εξακολουθούν να συζητούνται οι κανόνε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Με συνεργασία είμαι πεπισμένο ότι στο μέλλον νέοι κανόνε για το ποινικό δίκαιο θα θεσπίζονται μόνο όταν είναι απόλυτα αναγκαίο και ε, θα, οι αλλαγέ θα οδηγούν σε ποιοτική βελτίωση. Λοιπόν, αλλάξαμε τώρα. Πάμε στην διαδικασία προσέγγιση προσοχή του Προέδρου. Ο κύριο Λούαν δεν είναι παρόν και το λόγο δίνουμε στον κύριο Βό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κονέλη Δεγιόνγκ για την ε, δέσμευση που έχει αναλάβει και για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Είναι πολύ ισορροπημένο το κείμενο της έκθεσής του. Και βλέπω ότι ε, προτείνονται μικρά βήματα να πλησιάσουμε το συνολικό μας ε, στόχο. Χαίρομαι που βλέπω ότι σε κάθε κράτος μέλος το ποινικό δίκαιο έχει εξελιχθεί διαφορετικά και επομένως χρειαζόμαστε και διαφορετικά μέτρα εναρμόνισης και προσέγγισης χωρίς να περικόπτεται καμία θεμελιώδης ελευθερία. Χρειάζεται να προχωρήσουμε προσεκτικά και σε θέματα διαδικασίας και σε θέματα ουσιαστικού δικαίου. δεν ε, ε, θα έρθουμε σε σύγκρουση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασία Δεδομένων ούτε με καμία άλλη αρχή. Φοβούμαι ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να αναπτύξω περισσότερο αυτά τα επιχειρήματα. Πάντως ε, προτείνω να ακολουθήσουμε μια συνεπή διαδικασία και να μην, κάνουμε, να μην ξεκινήσουμε από το τέλος προς την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μάλμστρομ, θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω την ίδια γραμμή όπως και ο κύριος Φως. Πιστεύω ότι είναι επίγον να επωφεληθούμε της έκθεσης του κυρίου Ντεγιόν και να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια συντονισμένη στρατηγική για το πώς θα διαμορφωθεί το ποινικό δίκαιο και πώς θα το εναρμονίσουμε, ούτως ώστε να μην μπούμε σε τομείς όπου υπάρχουν βραχυπρόθεσμα ενδιαφέροντα, αλλά να εξετάσουμε και τους μακροπρόθεσμους στόχους για να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό ποινικό σύστημα δικαίου. Και με τους συναδέλφους από τον τομέα θεμάτων δικαιοσύνης θα μπορούσατε να συνεργαστείτε για να μπορέσουμε ε, να έχουμε κοινέ ε, προσεγγίσεις. Ε, αυτή είναι η προοπτική προς την οποία πρέπει να κινηθούμε και ξέρω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην προσέγγιση της οπτικής γωνίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παίξει ένα ρόλο μεσολάβησης και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το φροντίσετε. Ο κύριος Μπάτεν. Ε, Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει αυτά που για τα οποία προειδοποίησα του ε, εκλογεί μου στο Λονδίνο και του Βρετανού επί σειρά ετών. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να δημιουργήσει το δικό τη σύστημα ποινικού δικαίου. Αυτό το πρόγραμμα ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι πληρέστατο. Και το έγραψα σε μια δική μου έκθεση. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι δημιούργημα ευρωπαϊκή αστυνομία, αστυνομικού κράτου ευρωπαϊκού. Δεν χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στην Ευρώπη. Έχουμε το κοινό νόμο που χρειάστηκε, ε, η common law που χρειάστηκε χίλια χρόνια για να αναπτυχθεί στη χώρα μου. Έχουμε ρήτε διαφύλαξη, οι οποίε σαρώνονται από το νέο σύστημα και τη Magna Carta, τη Χάρτα Δικαιωμάτων και το Habeas Corpus Όλα αυτά έχουν παραμεριστεί. Ένα Βρετανό πολίτη τώρα μπορεί να αποσταλεί σε αδίποτε γωνιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα χαρτί, με αόριστε κατηγορίε και μπορεί να φυλακιστεί επί μήνε ή και χρόνια ακόμα. Τα βρετανικά και σκοτικά δικαστήρια, τα αγγλικά και βρετανικά τα σκοτικά και τα αγγλικά δικαστήρια επεμπόρισαν δικαιώματα του προστατεύσουν του πολίτε. Το δικό σα σύστημα θα κάνει για τι ελευθερίε αυτό που έκανε το νέο νόμισμα για την οικονομία σα, για τι οικονομίε σα. Ευχαριστώ κύριε Μπάτεν. Ο κύριος Πιχκέχ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ασχολούμεθα με το θέμα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο ώστε να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Με αυτή την έκθεση περνάμε απευθείας στη διαμόρφωση των στόχων. Γνωρίζουμε τη στρατηγική ε, της Επιτρόπου κυρίας Μάλμστρομ. Αν δεν ε, καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική και να έχουμε κάτι παράλληλα με το ποινικό δίκαιο στην Ευρώπη, τότε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία και οποιαδήποτε άλλη στρατηγική δεν θα έχει πραγματική ε, οντότητα υπό αυτή την οπτική γωνία εξετάζουμε την αρμόνιση του ποινικού δικαίου ευθυγραμμισμένο με τις εθνικές παραδόσεις και δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε μέσω του ποινικού δικαίου αυτό το οποίο ε, θα έπρεπε να κάνουμε μέσω της πολιτικής μας για την προστασία των συνόρων και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στο διαδίκτυο. Ε. Ο κύριος Πάσκα, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι οι συνθήκες ορίζουν ορισμένους τομείς και εδώ θα πρέπει να δούμε και το θέμα του ποινικού δικαίου και της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής για το ποινικό δίκαιο. Υπάρχουν ε, πολλές και διαφορετικές παραδόσεις ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Και ένας Βρετανός συνάδελφος ε, το εξέφρασε σαφέστατα και συμφωνώ ότι το Βρετανικό δίκαιο ε, ακολουθεί μια διαφορετική αντιμετώπιση από το δίκαιο των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μου έχουμε σαν βάση το αυστροουγγρικό δίκαιο και σίγουρα και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό οδηγεί σε διαφορετική στάση και αντιμετώπιση και γι' αυτό έχω αρκετούς δισταγμούς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε την πρωτοβουλία να εκπονήσει έκθεση για αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται τέλεια και με την ανακοίνωση που δημοσίευσε η Κομισιόν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Χαίρομαι που ουσιαστικά πέτυχε το στόχο της γιατί δρομολόγησε συζήτηση εντός και εκτός των θεσμικών οργάνων. Για πρώτη φορά είχα συνοψίσει ε, τις αρχές που διέπουν την νομοθεσία για το ποινικό δίκαιο ώστε να ενισχυθούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο νέο πλαίσιο της συνδίκης της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι ο στόχος αυτός ε, διαπνέει και τη δική σας έκθεση συμφωνούμε με την άποψη του εισηγητή ότι οποιαδήποτε νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σέβεται πλήρω τι αρχέ τη επικουρικότητα ε, και τη αναλογικότητα. Γνωρίζουμε βέβαια και έχει συζητηθεί ε, ξεκάθαρα και εδώ ότι υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές μεταξύ των κράτων μελών. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων που εγγυά το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για κάθε ε, για την νομοθεσία και το ποινικό δικαίωμα των ε, κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε πώς βέβαια μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Αλλά να έχουμε βέβαια κατά νου τις διαφορές και τις παραδόσεις στα νομικά συστήματα των διαφορών χωρών. Για την ενίσχυση λοιπόν των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προσπάθειες απαιτούνται σε συγκεκριμένους τομείς, θα παράσχουν όμως σημαντική προσθέμενη αξία. Είναι κάτι που είδαμε για παράδειγμα στα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Το 2008 και το 2009 θετήθηκαν δύο πολύ ε, σημαντικά μέσα, τα ε, πρώτα τα οποία εγκρίθηκαν με την κανονική ε, νομοθετική διαδικασία στον τομέα του ποινικού δικαίου. Υπήρξε πολύ επιτυχημένη συνεργασία των θεσμικών οργάνων και αυτό αποτελεί ένα καλό προηγούμενο και θα ελπίζουμε να επαναληφθεί και στο μέλλον. Θα δούμε επίσης ε, το insider dealing και την ε, χειραγώγηση των αγορών, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ε, και πρέπει να δώσουμε, για να το πετύχουμε αυτό, ένα μήνυμα ισχυρό ότι οι κοινοί κανόνες γίνονται σεβαστοί. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή τώρα των ποινικών μέτρων. Υπάρχουν με τη συνθήκη 10 εγκλήματα, 10 αξιόπινες πράξεις που ορίζονται ε, και θα πρέπει να ε, υπάρχουν οι κοινοί κανόνες και κοινοί ορισμοί. Έχουν γίνει πολλά μετά την Λισαβόνα. Εγκρίθηκαν οδηγίες ε, για την καταπολέμηση της οματεμπορίας, για την καταπολέμηση επίσης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και ολοκληρώνουν τη διαδικασία και για την οδηγία για το κυβερνό έγκλημα. Και θα έχουμε και μια νέα πρόταση για του νόμου περί κατασχέσεων. Είναι κάτι το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά έχουν συνεισφέρει στην ανάπτυξη ε, διατάξεων που θα οδηγήσουν σε μια ρεαλιστική ερμηνεία ε, μιας δέσμης κοινών κανόνων που θα είναι και ένα σημαντικό σημείο αναφορά για την περαιτέρω ανάπτυξη τη νομοθεσία νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ό,τι αφορά τα ποινικά ζητήματα. Βέβαια θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προβληματισμό και συζήτηση των νομικών ζητημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκροτήσει και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τον Ιούνιο και θα σα αναφέρω τα σχετικά από εργασία αυτή αυτής της διότι απαρτίζεται από, ε, από άτομα που έχουν ε, εμπειρία και γνώση, είναι επαγγελματίε του κλάδου, είναι νομομαθείς και σίγουρα θα κάνουν πολύ σημαντικές προτάσεις. Το ψήφισμα επίσης περιλαμβάνει πολύ σωστές προτάσεις. Μεταξύ αυτών να έχουμε μια απλούστερη γλώσσα ώστε και οι νομοθέτες ε, να καθοδηγούνται όταν θα πρέπει να συντάξουν κάποιες διατάξεις. Η ανακοίνωση περσινή της Κομισιόν αλλά και η έκθεση που συζητούμε σήμερα και που φαίνεται ότι έτυχε ευρείας υποστήριξη είναι μια αφετηρία ε, για τη χάραξη κοινή πολιτική στον τομέα του ποινικού δικαίου. Και περιμένω ε, να προχωρήσουμε μαζί με το Κοινοβούλιο ε, για ε, να επιτύχουμε πραγματικά έναν χώρο ασφάλειας δικαιοσύνης και ελευθερίας. Επόμενο σημείο, λέει πρόεδρος, είναι η έκθεση Μπόσκουρτ την κατάσταση της Τουρκίας, των γυναικών στη Τουρκία με προοπτική το 2020. Η συγκήτρια έχει το λόγο για 4 λεπτά.